Ναι, η ενίσχυση του συντονισμού και της μακροπροληπτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και θα βοηθήσει και το Συμβούλιο να ε, διεξάγει πλήρως τα καθήκοντά του. Ευχαριστώ ε, πολύ γιατί στην γνωμοδότησή μου καταφέραμε να συμπεριλάβουμε αυτές τις πτυχές η στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τη δυνατότητα του Συμβουλίου να ε, εντοπίσει σωστά, να αναλύει και να παρακολουθεί ε, πανευρωπαϊκούς συστημικούς κινδύνους η αυτονομία και η προβολή του Συμβουλίου ε, πρέπει να προστατεύονται ανα πάσα στιγμή. Σε αυτά τα πλαίσια η λογοδοσία, η διαφάνεια και η ανεξαρτησία του Συμβουλίου θα πρέπει να εγγυάται ε, και σε αυτό το πλαίσιο τα καθήκοντα της γραμματείας ε, του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι κατά, απόλυτα σαφή. Ο διορισμός του επικεφαλής ε, της γραμματείας θα πρέπει να γίνεται μετά από μια ανοιχτή και διάφανη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα ενημερώνονται ε, με επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας και φυσικά ο πρώτος αντιπρόεδρος θα πρέπει να διορίζεται με διάφορο τρόπο μέσω συμφωνίας μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωζώνης και σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια θητεία πέντε ετών διότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ισορροπημένη και αποτελεσματική εκπροσώπηση των κρατών μελών συνολικά. Η ε, διαχείριση και η σύνθεση του Συμβουλίου θα πρέπει να σέβεται το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς επίσης και την κυριαρχία των κρατών. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η δημοκρατία είναι απαραίτητες αρχές για να υπάρχει μια βιώσιμη και αξιόπιστη ε, χρηματοπιστωτική λειτουργία του συστήματος, εάν όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ε, προλάβει ή να μετριάσει αποτελεσματικά τους συστημικούς κινδύνους και να εγγυηθεί μια συνεκτική και δίκαιη ανάπτυξη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισήγητη για το σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο και υποστηρίζω θερμά. Το έργο σας ε, για την εξασφάλιση της διαφάνειας ε, είναι κάτι που η Άλντε πάντοτε θα υποστηρίζει. Δηλαδή αποτελεσματικό ε, συμβούλιο, συστημικό κίνδυνο αυτονομία, αφήνεια, αποτελεσματικότητα. Σημαντικοί παράγοντες. Αν θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα εντός ευρωζώνης, αλλά και στις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, έχω δύο ερωτήσεις προς τον εισηγητή. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί στο 10 και 12 διαγράφεται τον πρόεδρο του ε, Οπτικού Συμβουλίου και δεύτερο ερώτημα, αν κατάλαβα καλά η ΕΚΟΝ θα ψηφίσει τέλη Σεπτεμβρίου. Γιατί εμείς έχουμε προθεσμία κατάσταση τροπολογιών που λήγει την Πέμπτη, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο είχαμε για να εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήταν δυνατόν να αναβληθεί ίσως για την επόμενη εβδομάδα η λήξη της προθεσμίας. Όπως και αν έχει, ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρυσόγονο για το σχέδιο γνωμοδότησης. Εκπροσωπώ την Εύελιν Ρέγκνερ, άρα εκφράζω και τη δική της υποστήριξη στις προσπάθειες για διαφάνεια ανεξαρτής αυτονομία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδυνού. Η Εύελιν θα ήθελε να αναφερθούν κάποια περαιτέρω σημεία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το κείμενο. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του, του Συμβουλίου θα ήθελε η Εύελιν η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Συμβούλιο να ενισχυθεί, διότι κατά αυτήν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η επίβλεψη των μικροοικονομικών ανισορροπιών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τη συμμετοχή των σχετικών ε, εταίρων στις διαβουλεύσεις του Συμβουλίου οι φυγόμενε ομάδε, οι ομάδε που είναι σε κίνδυνο σε περίπτωση χρηματοπιστωτική κρίση, πρέπει να συμμετέχουν και ιδίω οι εκπρόσωποι των συνδικάτων αλλά και των ενώσεων καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν να είναι μέλη του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ως αντιστάθμιση, ως αντίβαρο. Και σε ό,τι αφορά τώρα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να ενισχυθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι και ο στόχος βέβαια του σχέδιου γνωμοδότησης, το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να έχει τις ίδιες εξουσίες, αρμοδιότητες με Κομισιόν και Συμβούλιο. Και ιδίω θα πρέπει να είναι σε θέση να εντέλεται ε, ελέγχους. Και κάτι τελευταίο, εξίσου σημαντικό όμως, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε αυτό το Συμβούλιο το εποπτικό. Κάτι δύσκολο ομολογούμε βέβαια, αν μόνο οι διοικητέ των κεντρικών τραπεζών είναι πρόσωποι που είναι άντρε στην πλειοψηφία του. Αλλά λοιπόν, παρόλα αυτά θα έπρεπε να επιμείνουμε στην διάσταση τη ισότητα των φίλων, στην ίση προσώπηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Επομένω. κατά κατάσταση τροπολογιών είχε οριστεί για την 22η Μαΐου. Αλλά μπορεί να παραταθεί, αν ζητηθεί, όπως ζητήθηκε δηλαδή κιόλας. 29 Μαΐου, μία εβδομάδα ακόμη, Ωραία. Μία παραπάνω εβδομάδα λοιπόν, 29 Μαΐου, 12 το μεσημέρι θα λήξει προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι εδώ ο κύριος ή δεν είναι. We continue. Δεν είναι ο κύριος Άγερ, θα πάμε στο 17. Προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης ε, για μια ακόμη φορά συντάκτη είναι ο κ. Χρυσόγονος, το οποίο στον οποίο δίνω και αλλού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι επιχειρήσει επενδύσεων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο γιατί διευκολύνουν ε, και οικονομίε ε, και τη ροή επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορε υπηρεσίε που χρησιμοποιούνται για να στηριχθεί η διαχείριση κινδύνων και κατανομή του κεφαλαίου. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα ισχυρό σύστημα προληπτική εποπτεία ε, ω προπόθεση στα αριθμιστικά συστήματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν λοιπόν έτσι να παρέχουν τι υπηρεσίε του πιο αποτελεσματικά στην Ένωση. Τα καθεστώτα που ισχύουν στην Ένωση ε, βασίζονται Ε, στην εφαρμογή των εθνικών ρυθμιστικών προτύπων ε, που ισχύουν για τους τραπεζικούς ομίλους, αλλά δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τους ειδικού κινδύνους ε, που είναι εγγενείς στις διαφορετικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων επενδύσεων. Η ισχύουσα, μάλλον η τρέχουσα πρόταση οδηγία στόχο έχει να αντιμετωπίσει τα τροτά σημεία και τους κινδύνους που είναι εγγενείς στις επιχειρήσεις επενδύσεων με Διακανονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προληπτική εποπτεία. Έχω καταθέσει λοιπόν τροπολογίε στο σχέδιο γνωμοδότησή με στόχο να τονίσουμε τι εξή βασικέ πτυχέ. Πρώτα απ' όλα, να ενισχύσουμε τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τι υποχρεώσει υποβολή αναφορών των επιχειρήσεων επενδύσεων στι εποπτικέ αρχέ μεταξύ των και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Το δεύτερο είναι να έχουμε πιο αυστηρές ακυρώσεις και πρόστιμα τα επιβάλλονται στις εν λόγω επιχειρήσεις από τις αρχές εφόσον αυτές δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Πιο συγκεκριμένα προτείνω να ενισχυθεί ε, ο αποτρεπτικός χαρακτήρας ε, των κυρώσεων, δηλαδή αύξηση των οικονομικών προστήμων αφενός, αλλά επιβολή στις ε, καταδικαστήσεις εταιρείε αφετέρου να δημοσιοποιούν τις κυρώσεις που τις επιβλήθησαν στην δική τους σελίδα και όχι μόνο στον ιστότοπο της ε, αρμόδιας εποπτικής αρχής. Ε, τρίτον, κατέθεσα κάποιες τροπολογίες που στόχο έχουν την καλύτερη ρύθμιση της πολιτικής απολαβών ε, και εποπτείας, παραδείγματος χάρη, περιορίζοντας το κειμενόμενο τμήμα στο 50% του πάγιου. Μιλάω για την απολαβή, για την αμοιβή. Και ένα άλλο σημαντικό είναι το άρθρο 29 της πρότασης. Θεωρώ ότι μια εταιρεία επενδύσεων που δέχεται έκτακτη οικονομική υποστήριξη δεν θα πρέπει να μπορεί ε, να ε, πληρώσει ε, κειμενόμενη αποδοχή. Να καταβάλει τέτοιου είδους αμοιβέ. Περιμένω και τις δικές σας παρατηρήσεις τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι σε γενικέ γραμμές βεβαίως δουλεύουμε πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ τεχνικός ο φάκελος. Επομένως, νομίζω προσυπογράφουμε τους στόχους. Χρειαζόμαστε ισχυρές κεφαλαγορές για να προωθήσουμε τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν ώψη του Brexit θέλουμε να προσελκύσουμε επενδυτικά κεφάλαια και ταμεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πρόσφατα είπε ότι οι επενδυτικές εταιρείες που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ελέγχουν το 80% των στοιχείων ενεργητικού του συνόλου των επενδυτικών εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι οι επενδυτικές εταιρείες είναι διαφορετικά πιστοτικά ιδρύματα, δεν είναι ακριβώς τράπεζες και λειτουργούν ανταγωνιστικά με τις τράπεζες διότι προσφέρουν επενδύσεις. Αλλά δεν δίνουν δάνεια και δεν δέχονται καταθέσεις. Διαχειρίζονται κεφάλαια, έχουν διαφορετικά επιχειρηματικά προφίλ και προς το παρόν λοιπόν πολλές από αυτές υπόκεινται σε νομικές εξαιρέσεις βάσει εθνικής νομοθεσίας. Και όλα αυτά πλήττουν τη λειτουργία αυτό το συγκεκριμένο πλήττει τη λειτουργία και την ακαιρεότητα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διακρίνει 11 κατηγορίες επενδυτικών εταιριών και η πρόταση αφορά μόνο τις τρεις. Τις πολύ μεγάλες συστημικές επενδυτικές εταιρίες, οι οποίες ε, κατατάσσονται στην κατηγορία 1 και παραμένουν στο CRS-EAD, δηλαδή πολύ αυστηρό έλεγχος συστημικός βάσει των οδηγιών και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία 2 είναι λιγότερο συστημικές οι επενδυτικές εταιρείες, αλλά πρέπει να πληρούν τα, τις προδιαγραφές. Ε, κατηγορία 3 είναι οι μικρές επενδυτικές εταιρείες και δεν υπάρχει υποχρέωση να έχουν κεφαλαϊκή επάρκεια με συγκεκριμένα προαπαιτούμενα κεφαλαϊκής επάρκειας όπως η κατηγορία 1 και 2 συμμερίζομαι τις απόψεις του εισηγητή σε μεγάλο βαθμό οι ενισχυμένες κυρώσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνώ για αυτό. Πρέπει να το ελέγξω ότι δεν είναι υπερβολικά υψηλές κυρώσεις. Νομίζω ότι η διατύπωση είναι πραγματικά ε, πολύ ισχυρή. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα πρόστιμα. Και υπάρχει και το θέμα των αμοιβών. Πρέπει να δούμε εάν οι αμοιβέ έχουν να κάνουν με αυτούς που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο, με τους εμπλεκόμενους φορείς σε αυτές τις τρεις κατηγορίες επενδυτικών εταιριών ή αν μιλάμε μόνο για συγκεκριμένα επενδυτικά ε, κεφάλαια ή ταμεία. Θα ήθελα ο εισηγητής να μου δώσει λίγο χρόνο να τα ελέγξω αυτά. Ευχαριστώ. For uh, uh, Επίσης, μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει αύριο και ο εισηγητή στην εικόνα, αφού θα γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων εκεί, θέλει να προχωρήσουμε γρήγορα. Αλλά δεν ξέρω αν θα περάσει το θέμα από την εικόνα, γιατί χρειάζονται πολλά περισσότερα στοιχεία για τα διάφορα είδη επενδυτικών εταιριών. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να πάρει το λόγο κάποια στιγμή για αυτό το θέμα. Βλέπω πως όχι. Άρα καταλεκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 29 του μηνός στις 12 το μεσημέρι. Η κυρία Ντελβό και ίσως λίγο αργότερα, αν μπορεί να γίνει αυτό, λίγο αργότερα παρακαλώ. Καλώς. Η γραμματεία θα το δει κατά πόσο μπορεί να είναι αυτό. Ε, το κρατάμε για τις 29 Μαΐου και αν μπορέσει η γραμματεία θα το παρατείνει. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Ντελβό, και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Προχωρούμε στο σημείο 18 της ημερήσιας διάταξη. Εξέταση του εφαρμοστέου δικαίου στα αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων έναντι τρίτων. Και εγώ είμαι εισηγητή. Να σας πω κάποια βασικά στοιχεία. Δυστυχώς η έκθεση είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά προς το παρόν. Ελπίζω όμως θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πάρα αυτά. Και ε, διότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει να αποτελείται από 15 άρθρα και ε, ακολουθεί στενά τους κανονισμούς ROM 1 και ROM 2. Γι' αυτό και εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο στα άρθρα που ε, ε, βρίσκονται σε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόνο. Και δεν ασχολούμαστε με τα άρθρα που υπάρχουν κι αλλού, που έχουν απλά αντιγραφή από τους δύο προηγούμενους κανονισμούς που ανέφερα. Ως προς το βασικό για ε, το εφαρμοστέο δίκαιο, το σχέδιο ε, έκθεση ζητά ο νόμος της συνήθους κατοικίας του εκχωρούντος να ισχύσει γιατί έχουν ψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και προβλεψιμότητας με αυτόν τον τρόπο. Είναι, ε, επίσης προτείνεται μάλλον οι εκχωρήσεις που γίνονται στο πλαίσιο συλλογικών διαδικασιών να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του προτινόμενου κανονισμού. Ο κανονισμός 2015 κάθετος 8.4.8 για τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας ήδη περιλαμβάνει κανόνες και διατάξεις για το θέμα της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Το σχέδιο έκθεσης ε, αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι συνέπειες έναντι τρίτων για τους οφειλέτες ε, ρυθμίζονται μόνο από τον κανονισμό ΡΟΜ 1. Άρα μας ζητά να αποκλείσουμε ρητά ε, ε, αυτά τα τρίτα μέρη με βάση την προτινόμενη νομοθεσία. Από την προτινόμενη νομοθεσία. Αυτά είναι τα βασικά. Το περιεχόμενα της εισήγησης, της έκθεσης. Έχετε το λόγο, η κυρία Ντελβό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επομένως, κοιτάξτε, διάβασα την πρόταση και νομίζω ότι δεν είμαι βέβαια ειδικό, αλλά νομίζω ότι πράγματι δείχνει η Επιτροπή μια ισχυρή βούληση να δημιουργήσει ένα αρμονισμένο νομικό πλαίσιο και έχει στόχο να ενισχύσει την νομική ασφάλεια έτσι περαιτέρω. Παρόλο που ε, λυπούμε πολύ για το γεγονός ότι αν δεν απατώμε, καμία οργάνωση καταναλωτών δεν συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση. Θα ήταν ενδιαφέρον για εμάς να είχαμε την άποψή τους και τη γνώμη τους. Έχω κάποιες ερωτήσεις περισσότερο παρά σχόλια να υποβάλω. Κύριε Πρόεδρε, εσείς ως εισηγητής, προτείνετε να αποκλειστεί ο φιλέτης από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή. Μήπως υπάρχει σύγκρουση νομοθεσίας μεταξύ του σχεδίου αυτού και του άρθρου 14.1 του κανονισμού ΡΟΜ 1 Πρώτη ερώτηση αυτή. Και δεύτερο, για την τρίτη τροπολογία που διευρύνει το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού και συμπεριλαμβάνει την μεταβίβαση, την εκχώρηση των συμβάσεων. Καλά κατάλαβα δηλαδή ότι αποκλείεται η εφαρμογή του κανονισμού ΡΟΜ 1 για το ζήτημα αυτό. Τρίτο ερώτημα, για την τιτλοποίηση ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή προβλέπει εξαίρεση για τις συμφωνίες τιτλοποίησης και γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου και θα ήθελα πραγματικά να μου δοθούν απαντήσεις. Ευχαριστώ. Uh, does the Commission wish to take the floor on that? Θέλει η Επιτροπή το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μόλις έφτασα και μόνο το τελευταίο ερώτημα άκουσα. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ. Ναι, το τελευταίο ερώτημα είχε να κάνει με την τίτλοποίηση γιατί προβλέπεται εξαίρεση για τις συμφωνίες τίτλοποίησης και γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με την πρόταση του εισηγητή να αποκλειστούν οι οφειλέτες από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κανονισμού. Υπάρχει ε, ε, το άρθρο 14 του ΡΟΜ 1 αντίκειται στην ουσία αυτού του κανονισμού. Μήπως υπάρχει σύγκρουση εκεί νομική και μετά. Τρίτο ερώτημα. Συμπεριλαμβάνονται, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογή γιατί συμπεριλαμβάνεται η εκχώρηση των συμβάσεων. Άρα αποκλείεται η εφαρμογή του ΡΟΜ 1 πάνω σε αυτό το σημείο. Έτσι δεν είναι. Αυτό θέλετε να κάνετε, αυτό, αυτός είναι ο σκοπός μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, οφείλω να πω ότι δεν είμαι σε θέση, δεν, δεν, έχω, δεν μπόρεσα να διαβάσω την έκθεση, δεν την βρήκα πουθενά. Άρα δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα για τον αποκλεισμό του οφειλέτη, γιατί δεν έχω διαβάσει την έκθεση, δεν μπορούσα να τη βρω πουθενά. Θα προσπαθήσω να σας δείξω τη θέση μας για τις άλλες δύο ερωτήσεις σας, για την τιτλοποίηση, γιατί να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση αυτή έχει να κάνει με, με τρίτα μέρη. Άρα, ο νόμος της συνήθους κατοικίας του εκχωρητή, του εκχωρούντος, πρέπει να είναι ο νόμος που ισχύει, σε σχέση με τις δύο άλλες δυνατότητες οι οποίες βασίζονται στην αυτονομία των μερών. Δεν το, ε, τα συμβαλόμενα μέρη δεν τα έχουν διαλέξει ως ε, νομική ισχύ και γι' αυτό ε, μιλούμε για τη συνήθη κατοικία, αυτού που εκχωρεί. Όμως προσκρούσαμε σε πολύ ισχυρή αντίθεση από τους συναδέλφους που ασχολούνται με τις χρηματαγορές. Δεν το θέλουν αυτό. Η τιτλοποίηση αυτή τη στιγμή, το securitization, γίνεται από πολύ μεγάλους φορείς, πολύ μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολύ μεγάλες τράπεζες, οι οποίες είναι σε θέση να δομήσουν και να διαρθρώσουν αυτά τα τμήματα τιτλοποίησης και συναλλαγών τέτοιου είδους με τρόπο ώστε να ισχύει ο πιο ευνοϊκός νόμος για το τρίτο ε, μέρος και να είναι ο νόμος εκεί όπου υπάρχει η διεκδίκηση, η, ε, η εκχώρηση έναντι τρίτων. Δηλαδή, συμφωνούν όλοι αυτοί με τους οφειλέτες ότι αρμόζει και ταιριάζει καλύτερα να ομαδοποιηθούν οι εκχωρήσεις έναντι τρίτων, αναλόγως με την νομοθεσία που ισχύει για το περιεχόμενο κάθε μίας. Άρα δομούν τις συναλλαγές έτσι ώστε όλες οι διεκδικήσεις που ε, εκχωρούνται να διέπονται από το ίδιο δίκαιο. Δηλαδή ομαδοποιούν αυτά τα προϊόντα με βάση ε, έτσι ώστε να υπάγονται όλα στο ίδιο δίκαιο σε κάθε ομάδα, τα μέλη της ομάδας, τα μέλη του πακέτου αν θέλετε. Άρα η Επιτροπή μπορεί να διαλέξει ή να υποβάλει πρόταση ή να μην υποβάλει καθόλου πρόταση γιατί οι χρηματαγορές ε, τα στήλωσαν και είχαν μια πραγματικά αδυσόπιτη και πολύ στεναρή αντίδραση. Και είπαμε λοιπόν ότι να έχουμε τη συνήθεια κατοικία αλλά τα συμβαλόμενα μέρη που ασχολούνται με την τιτλοποίηση να τα διαλέξουν τα ίδια, άμα θέλουν να διατηρηθεί ο νόμος της συνήθους κατοικίας ή αν θέλουν κάποιο άλλο δίκαιο να ισχύσει. Δηλαδή, σεβόμαστε τις πρακτικές και τα έθιμα των μεγάλων τραπεζών και των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά επιτρέπουμε και στους μικρότερους να μπουν στην αγορά της τιτλοποίησης, γιατί τους επιτρέπουμε να υπαχθούν στην συνήθη νομοθεσία που είναι ε, να ισχύσει η νομοθεσία του συνήθους τόπου κατοικίας του εκχωρηθεί κτλ. Θεωρούμε ότι έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιώνει και τους μεν και τους δε, ε, είναι δίκαιη στην αντιμετώπιση υιοθετούμε το σύνηθες αυτό που εμείς θέλουμε και οι μεγάλες τράπεζες μπορούν να διατηρήσουν και αυτές τα συμφέροντά τους γιατί αυτές θέλουν να ομαδοποιούν τα προϊόντα και δεν θέλουν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαταράξει τις συνήθεις διαδικασίες ε, όσων κάνουν τιτλοποιήσεις και γι' αυτό διαλέξαμε ισορροπημένη λύση, δηλαδή ίδιος κανόνας για όλους, ο νόμος του, της συνήθους κατοικίας, εάν όμως το προϊόν είναι έτσι δομημένο, τότε τα συμβαλώμενα μέρη να διαλέξουν άλλο δίκαιο εάν το επιθυμούν. Είναι καλή συμβαστική λύση αυτή. Ίσως φαίνεται περίεργο η αυτονομία των μερών να είναι αυτή που θα διαλέξει το δίκαιο που θα ισχύσει έναντι των τρίτων, Φαίνεται κάπως περίεργο και ακούγεται περίεργο αυτό, αλλά είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Τώρα για την εκχώρηση ή μεταβίβαση των συμβάσεων. Αυτό έχει γύρει ορισμένες αμφιβολίες. Η πρόταση αυτή δεν καλύπτει αυτή την περίπτωση. Η πρόταση αυτή αναφέρει αυτό το θέμα μόνο στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ του δικαιούχου και αυτού στον οποίο εκχωρήθηκε η σύμβαση. Είναι σημαντικό να αποφασίσουμε ποιο δίκαιο θα ισχύσει για το ποια ένομα συμφέροντα έχουν προτεραιότητα εναντί των άλλων Εάν έχουμε μια κανονική εκχώρηση μιας διεκδίκησης και στη συνέχεια αυτή μεταβιβαστεί μέσα σε μια σύμβαση, αυτό συμβαίνει. Η αγορά, οι τράπεζες, κατά τύχη, από ατύχημα, η ασκεμένα, εν πάση πτώση, είναι πράγματα που συμβαίνουν πολύ συχνά και μπορεί να υπάρξει ε, διαφωνία για την προτεραιότητα σε ό,τι αφορά το δικαιούχο και αυτόν στον οποίο έχει εκχωρηθεί η σύμβαση. Και γι' αυτό λέμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τις εκχωρήσεις έναντι τρίτων. Όμως δεν παρεμβαίνουμε στη μεταβίβαση των συμβάσεων ή στην εκχώρηση αυτών. Δεν αποφασίζουμε το εφαρμοστέο δίκαιο για το trading, για το clearing ή για το settling, για την εκαθάριση των λογαριασμών και όλα αυτών συναλλαγών. Όλα αυτά ε, ε, πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες της χρηματαγοράς που να μην προβλέπουν διακρισιακή ή διακριτική μεταχείριση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, η κυρία Ντελφό, πήρατε τις απαντήσεις που θέλετε, γιατί θα ήθελα να προσθέσω κάτι για την τροπολογία 3, η οποία έχει ως στόχο την αιτιολογική σκέψη να την κάνει να την πλησιάσει τις υλικές διατάξεις, τις ουσιώδεις διατάξεις όπως τις προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η τροπολογία 13 ο σκοπός της αλλαγής αυτής είναι το εφαρμοστέο δίκαιο να πλησιάσει περισσότερο τις εκχωρήσεις. Τις εκχωρούμενες απαιτήσεις. Άλλα σχόλια υπάρχουν. Προτινόμενη καταληκτική προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 24η Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λογικά θα συνεχίσουμε με το άρθρο 20, ε, με το σημείο 20, αλλά δεν είναι εδώ οι εισηγητές, η κυρία Κέπχαρ και ο κύριος ε, Φως, για τις συμβάσεις παροχής ε, ψηφιακού περιεχομένου. Πρέπει να το αναβάλουμε λοιπόν το σημείο αυτό. Στη συνέχεια έχουμε το σημείο 21, την επικουρικότητα, που είναι κάτι για το οποίο λαμβάνεται γνώση. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο το οποίο είχαμε παραλείψει, το σημείο 14, ανταλλαγή απόψεων για τους κανόνες και τις γενικές αρχές που αφορούν μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη-μέλη ε, για την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε δύο επιλογές. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Σάγερ, ο οποίος δεν είναι εδώ αλλά έχω ε, την παρέμβασή του. Επομένως, αν θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω την παρέμβασή του ή θα περιμένουμε ένα τέταρτο να έρθει ο κύριος Σάιερ. Ε, εσείς αποφασίζετε να τα πω. Εντάξει. Εγώ ως Κύριε Σάγερ, θέλω να σας πω ότι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σχετική πρόταση αφορά το πλαίσιο της επιτροπολογίας και την υπόθεση της γλυφοσάτης. Βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ένα πολύ χαμηλό αριθμό περιπτώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα, η διαδικασία της επιτροπολογίας ε, ε, οδήγησε σε μία εκδοχή ε, χωρίς γνώμη και αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει κατά πόσον θα εγκρίνει την εκτελεστική πράξη ή ε, όχι. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους δεν υπάρχει γνώμη ε, ότι είναι πάρα πολύ λεπτή και επομένω προτείνει την εξή τροπολογία η οποία κατά την άποψή της θα επιτρέψει να αποφύγουμε τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει γνώμη. Οι τέσσερις τροπολογίες είναι οι εξή. Πρώτον, η δυνατότητα να υπάρχει περαιτέρω συνεδρίαση της Επιτροπής Εφέσεων σε ε, υπουργικό επίπεδο. Δεύτερον, προτινόμενη αλλαγή τη μεθοδολογίας των κανόνων ψηφοφορίας ε, στην Επιτροπή ε, προσφυγών και ε, επίσης συζήτηση των αποτελεσμάτων της αποκάλυψη συγγνώμη, των αποτελεσμάτων της ψηφοφορία. Ε, τέταρτον, η δυνατότητα να παραπέμπονται συγκεκριμένες περιπτώσεις σε περίπτωση που υπάρχει ε, απόφαση για μη γνώμη ε, για να δώσει η Επιτροπή Ενστάσεων μια μη δεσμευτική απόφαση προς το Συμβούλιο. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα πρέπει να εξετάσει τη λειτουργία της διαδικασίας επιτροπολογίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν λόγοι για την πρόταση, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η διαδικασία της επιτροπολογίας είναι αποδεδεγμένα ε, μια διαδικασία που λειτουργεί αποτελεσματικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεύτερον, θα εξετάσω τις τέσσερις συγκεκριμένες τροπολογίες και επίσης είναι καθήκον μου να αναφέρω ότι λάβαμε πέντε γνωμοδοτήσεις μέχρι τώρα από τις επιτροπές MV INTA, ΕΚΟΝ, ΙΤΡΕ και ΑΓΡΙ και ακόμα είμαστε εν αναμονή μιας ε, γνωμοδότησης από την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Ε, τρεις ε, βουλές κρατών μελών ε, γνωμοδότησαν επί του θέματος. Η Γαλλία, η Δημοκρατία και η Πολωνία και θα λάβουμε υπόψη και τις δικές τους γνωμοδοτήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του κυρίου Σάιερ. Σχόλια από τα μέλη, κυρία Κάουφμαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κρίμα που ο Τσανάλφος Σάγερ δεν μπορεί να είναι εδώ διότι εδώ και χρόνο ασχολείται εντατικά με το θέμα αυτό. Μπορώ όμως ε, να συμφωνήσω απόλυτα σε ό,τι αφορά την γλυφοζάτη που ε, καταδεικνύει με υποδειγματικό τρόπο, θα έλεγα, το ζήτημα. Τα κράτη-μέλη τελικά απεμπολούν τις ευθύνες τους ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που καλύτερα να βγάλει τα κάστανα με τη φωτιά. Και Υπάρχει αυτή η πρόταση της Κομισιόν ό,τι αφορά την εκτελεστική ε, πράξη για αλλαγή της διαδικασίας. Ε, θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό. Σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση τώρα ε, στην ΑΦΚΟ, συζητείτε, όπως είπατε ακόμη το θέμα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ψηφοφορίας προτείνονται δραστικές αλλαγές και μια ε, πρόταση για τους ε, υπουργούς ε, και είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία ψηφοφορίας των εκπροσώπων στις επιτροπές, στην Επιτροπή Προσφυγών. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ε, δυνατότητα οι πολίτες να παρακολουθούν ε, τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν αποφάσεις ε, οι εκπρόσωποι τους. Το θεωρώ ότι είναι σωστό λοιπόν να υπάρχει αυτή η δημόσια πρόσβαση. Δηλαδή να μην μιλάμε μόνο για τις Βρυξέλλες που αποφασίζουν, έχουν εθνικά πρόσωπα οι Βρυξέλλες και επηρεάζουν τις αποφάσεις και αυτοί. όπως για παράδειγμα το πρόβλημα της κλιφοζάτης και βιώσαμε όλοι μας ε, το θέμα αυτό. Ρόντε. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Αν δείτε τα όσα λέει το θέμα, είναι ιδιαίτερα τεχνικό, αλλά τρόπον την το θέμα αυτό πάντα επισημαίνει τις ομοιότητες ε, ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους πολίτες στα κράτη-μέλη ως Ευρωπαίους. Τα θεωρούν Γερμανούς, Δανούς, ε, Πολωνούς και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και για μένα είναι παράλογο να έχουμε ένα τόσο ανοιχτό κοινοβούλιο, ίσως είναι ένα από τα πιο ανοιχτά κοινοβούλια στον κόσμο, αλλά οι πολίτες στην Ευρώπη θεωρούν ότι το μόνο που κάνουμε στην Ευρώπη είναι και κλεισμένο των θερών, δεν υπάρχει καμία διαφάνεια και γιατί αυτό, γιατί το Συμβούλιο είναι απόλυτα κλειστό και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από πλευράς πολιτών και από πλευράς κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό και φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσά συμφωνείτε. Και αυτή η εξέταση της διαδικασίας με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Συμφωνώ με τον εισηγητή και τα όσα μας είπατε εσείς εκ μέρους του, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί νομίζω τα περισσότερα τα ανέφερε πολύ σωστά η κυρία Κάουφμαν. Και θα πω απλώς να προχωρήσουμε και να υποστηρίξουμε την πρόταση, αλλά να είναι μόνο η αρχή η όλη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω με την ιδιότητα του εισηγητή της ΑΦΚΟ, διότι είμαι εισηγητή στην Επιτροπή ΑΦΚΟ για τη γνωμοδότηση για το θέμα αυτό και να σας πω απλώς ότι έχουμε μια δυσκολία στη γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ. Ε, θα μπορούσε να είχε προχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά υπάρχει εξή δυσκολία. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μεγάλων πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου και δεν μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τη συμβαστική πρόταση, η οποία ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί. Να πω δηλαδή απλώ ότι στην Επιτροπή Σταγματικών Θεμάτων, όπω ακριβώ ακούστηκε προηγουμένω και από του συναδέλφου, εμεί υποστηρίζουμε σίγουρα την αρχή που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε διάφορες καταστάσεις. Το μόνο θέμα στο οποίο είμαι αντίθετο και είμαι αντίθετο φυσικά και εδώ και στην ΑΦΚΟ, είναι αν είναι όντως ευσεβής ο στόχος, τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας είναι τα καλύτερα το να πάμε λοιπόν σε τρίτο επίπεδο στους υπουργούς όταν το θέμα έχει ε, μπλοκαριστεί σε επίπεδο συμβούλων ε, θα βελτιώσει κάτι ή θα προσθέσει ένα ακόμα επίπεδο το οποίο δεν θα οδηγήσει πουθενά. Πιστεύω λοιπόν ότι με τον ίδιο στόχο με τον οποίο συμφωνώ θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε μια λύση η οποία να είναι λίγο πιο αποτελεσματική και αυτό σημαίνει ότι δεν θα αντικαταστήσουμε κάτι αυθαίρετο που είναι το Συμβούλιο με τον κίνδυνο μιας άλλης αυθαίρετης απόφασης ε, που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν ε, υπάρχει κατάλληλη πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, τα οποία αφορούν την υγεία, αφορούν ε, θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τους ανθρώπους και επομένως εάν δεν μπορεί να υπάρξει πλειοψηφία στο Συμβούλιο κανονικά δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να δώσει έγκριση για ένα προϊόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια δυναμία, ε, μια ανικανότητα να αποφασίσει κάποιο ε, και να δίνουμε τη δυνατότητα σε ένα τρίτο, σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αποφασίσει εκ μέρου των κρατών μελών. Είναι το μόνο σημείο στο οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Δεν είναι θέμα διάσταση απόψεων ως προς την αρχή, αλλά να μην δώσουμε τελικά την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετεί που δεν τις έχουν δώσει συνθήκες. Η Κομισιόν θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα θετικά σχόλια και την στήριξή σας. Μια πολύ σύντομη αντίδραση στην τελευταία παρατήρηση του κύριου Ντουράν για από την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Ναι, έχουμε σημειώσει το σχόλιο αυτό και ήδη συμμετείχαμε και στη συζήτηση στην Επιτροπή ΑΦΚΟ, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι φυσικά ότι αυτό αντιστρέφει τη λογική του κανονισμού της επιτροπολογίας που είναι ότι χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για να σταματήσει και να μην επιτρέψει την έγκριση μιας εκτελεστικής πράξης. Και αυτό φυσικά βαρύνει ε, ουσιαστικά τη διαδικασία της επιτροπολογίας και των εκτελεστικών πράξεων, δηλαδή την ομαλή εφαρμαγή της ε, βασικής νομικής πράξης τις επιλογές πολιτικής ε, τις ε, ε, ε, έχετε κάνει ήδη εσείς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Συνομοθέτες. Ε, και αυτό είναι στη βασική νομοθετική πράξη και δεν θα έπρεπε να επανερχόμαστε στο θέμα αυτό στη διαδικασία της επιτροπολογίας. Αυτό είναι η μόνη μας διαφωνία, αλλά κατά τα άλλα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα σχόλιά σας διότι μας στήριξαν. Ευχαριστώ. Το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι να ανακοινώσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 20 και 5η 21 Ιουνίου. Και αυτά για τη συνεδρίαση. Έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών στις 5 η ώρα. Παρακαλώ να είστε στην ώρα σας. Ξέρω ότι ο κύριος Φως ε, θα βιάζεται. Ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σε μια ώρα.